Αγαπητοί συνάδελφοι, τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα κείμενα που εγκρίθηκαν είναι στην διάθεσή σας. So, colleagues, the of yesterday's... Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι στη διάθεσή σας όπως είπα. Θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχουν σχόλια στα χτεσινά πρακτικά, εάν όχι εγκρίνονται. Περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου. Συνάδελφοι παρακαλώ. Ως συνήθως σας ζητάω να κάνετε λίγη ησυχία γιατί κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να μιλήσουν. Περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου. Ξεκινάμε με την έκθεση του κυρίου Λαντσμπέργης, ε, τελωνιακά, ε, τελωνιακή δασμή σε αγαθά προέλευσης Ουκρανίας. Ο κύριος Για Πέτερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πώς βοηθάει κανείς. Ναι, ναι, το ξέρω. Πώς βοηθάει κανείς μια χώρα που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, όπου βλέπουμε πως υπάρχει ο κίνδυνος μέσω αυτών των δυσκολιών να κινδυνεύσει ο δημοκρατικός μετασχηματισμός. Τη βοηθάμε αυτή τη χώρα με το να της δίνουμε το χέρι για οικονομικές σχέσεις. Και αυτό ακριβώς υπάρχει σε αυτή την ε, σε αυτό το ψήφισμα. Να δώσουμε δηλαδή τη δυνατότητα να έχει μια ευκαιρία να κάνει εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχετικές διευκολύνσεις. Και βεβαίως θα πρέπει να έχουμε αυτές τις ουσιαστικές σχέσεις και να τις διευκολύνουμε όπως ε, θεωρεί άλλωστε και η του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ντάνιελ Χάναν για ένα λεπτό. Χάναν. Ευχαριστώ. Εξεπλάγην από τον αριθμό των βουλευτών εδώ μέσα που είναι διατεθειμένοι να γίνουν υποχείρια του Πούτιν ενώ αυτοαποκαλούνται πατριώτες και εθνικιστές στις χώρες τους. Δηλαδή η λογική ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου έχει οδηγήσει τους ανθρώπους να υπερασπίζονται μια ιδεολογία και μια οργάνωση που είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, και εγώ θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια, ένας αντιδημοκρατικός εκβιασμός, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα της Ουκρανίας, θα να ζουν σε μια κανονική χώρα όπου τιμούν τα συμβόλαια, είναι ασφαλής ιδιοκτησία και μπορεί να στηρίξει κανείς αυτό το σύστημα είτε στηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι. Εγώ θέλω μια Ευρωπαϊκή Ένωση διεθνή, κοσμοπολίτικη και αισιόδοξη και καθόλου δεν μπορώ να συμπλέψω με τον πουτινισμό. Σας ευχαριστώ. Κύριο έχω εδώ πέρα στον κατάλογο. Then uh, give the floor to Mr. Luke. Luke. Ο κύριος Λούκε, έχει το λόγο λοιπόν εφόσον δεν είναι στην αίθουσα. Κυρία Πρόεδρε, δεν ψήφισα εγώ γιατί δεν μου αφήσατε να μιλήσω επί της διαδικασίας. Άρθρο 140 παράγραφος α του κανονισμού λέει πως το Κοινοβούλιο θα πρέπει να βλέπει τις οικονομικές επιπτώσεις των ε, νομικών του πράξεων. Εδώ πέρα δεν αναφέρονται οικονομικές επιπτώσεις. Δεν ήξεραν τι ψηφίζουν άρα οι βουλευτές. Η πρόταση της Κομισιόν δεν περιέχει νούμερα. Και το τι, ε, ποια θα είναι τα ε, έξοδα τα οποία θα έχουμε τι επίπτωση θα έχει το να μην επιβάλλουμε δασμούς. Έχω δικαίωμα να μιλήσω επί του κανονισμού το οποίο περιεκόψατε. Δεν ήταν σύνομο αυτό. Έχετε κάποιες υποχρεώσεις ως πρόεδρος και με εμποδίσατε να ενημερώσω το σώμα. Ότι λαμβάνει δηλαδή μια απόφαση χωρίς να ξέρει τις οικονομικές της επιπτώσεις. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην έκθεση Σάρβαμα για την απαλλαγή των Ευρωπαϊκών Φημιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Έτοιμα της κυρίας Μακλάρκιν για να πάρει το λόγο. Είναι μέσα στην αίθουσα. Όχι. Περνάμε λοιπόν στην έκθεση Deutsch απαλλαγή του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πάλι ο κύριος Πίτερ Γιάρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και χαίρομαι για το ότι το Κοινοβούλιο έλαβε μια απόφαση ε, να μην δώσει απαλλαγή. Είχαμε τη συζήτηση για τον προπολογισμό και ακόμα και εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο άμεσα θα ήθελα να παρακαλέσω το Συμβούλιο να πληρώσει στον προϋπολογισμό το υπόλοιπο των εισφορών των κρατών μελών. Δεν είναι δυνατόν να είναι μια χώρα κράτος μέλος και να μην πληρώνει στην ώρα της ε, αυτά τα οποία οφείλει στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι Σα Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Γιάρ. Εδώ έχει ολοκληρωθεί ο κατάλογος των ομιλητών και λίγη συνεδρίαση. Τα πρακτικά θα υποβληθούν στο Κοινοβουλίο προς έγκριση για την άρχιση επόμενη ε, Συνόδου Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ε, θα προωθήσω τα εγκεκριθέτα σήμερα ψηφίσματα στους αρμόδιους φορείς που αναφέρονται στα ψηφίσματα, διακόπτεται η συνεδρίαση.